Vous êtes bien bruyants, les collaborateurs, là. Allez. Le projet d'ordre du jour. Λοιπόν, το σχέδιο μέσα διάταξη μπορεί να εγκριθεί αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ανακοινώσει τη Προέδρου. σα δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, να κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε ποιοι είναι οι παρόντες και αν υπάρχει απαρτία. Άρχεται η ψηφοφορία. Je ferme le vote. Πέρα στις ψηφοφορίες. Λοιπόν, κυρία Σεύσκα δεν έχετε την κάρτα ψηφοφορίας, το σημειώνουμε. Θα ψηφίσετε ε, διαχειρός και έχουμε έναν σοσιαλιστή παραπάνω. Λοιπόν, άρα ε, διαλέξτε μεταξύ ε, των παρόντων ένας δεν θα ψηφίσει. Α, ωραία, τώρα έχουμε το σωστό αριθμό. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό 1008 του 2008 για τους κοινούς κανόνες για την εκμετάλλευση των ε, αεροπορικών υπηρεσιών στην κοινότητα της κυρίας Ταβαρντέλ. Θα ψηφίσουμε την διαπραγματευτική εντολή. Άρχεται ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. Η κυρία Λουκασέφσκα είναι υπέρ. Πέρας. Α, έχετε τελικά την ε, κάρτα σας. 35 υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κυρία Ταπαντέλ. Θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Αλλά μόλις ξεκινήσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την έκθεση Κριστίνου dallon για την επιβολή τελών, την οδηγία στα βαρέα οχήματα. Πρόταση οδηγίες για τη φορολόγηση των βαρέων φορτηγών που χρησιμοποιούν ορισμένες υποδομές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 208 υπέρ κατά άποχες Απορρίπτεται. 23 της ένβη υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές λοιπόν να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Λοιπόν, έχουμε τις 2.66, 3.63 και 198 που θα ψηφιστούν από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Είκοσι έξι. Υπέρ. Κατά άποχες. Λοιπόν, να ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά να ελέγξουμε. Άρχιτε προφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες, οι 2.21 και 26 της ένβη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 27 ένβη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λάθος. Η 226 καταπίπτει γιατί μόλις εγκρίναμε την 27. Συγγνώμη. Λοιπόν, δύο ταυτόσιμες, 227 και 28 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε και εδώ. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ελέγχουμε. Mm. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται με μία ψήφο πλειοψηφία. 2.62 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε άρχεται πέρας ναι ναι απορρίπτεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ε, καλά, ωραία, ελέγχουμε. Την συμβαστική 3. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 19 υπέρ, 19 κατά. Λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε μία-μία τις τροπολογίες τότε. Λοιπόν, μαζί 17 και 29. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε αυτές τις δύο ταυτόσημες άρχεται. Πέρας. Πέρας. 19, 19 απορρίπτονται. Άλλες δύο ταυτόσημες. 268 και 271. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές έλεγχος άρχεται περάς 19-19 απορρίπτονται λοιπόν 269 υπέρ παρακαλώ κατά άποχες έλεγχος πέρας απορρίπτεται 2.70 υπέρ παρακαλώ κύριε Βιμ Βαντεκόπ μην ενοχλείτε τον κύριο Μπάρτ σας βλέπω τόση ώρα, τόση ώρα σας κοιτάω. Λοιπόν, 2,70 έλεγα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίφθεται. 2,72 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίφθεται. 2,73 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4α υπέρ παρακαλώ κατά άποχες εγκρίνεστε συμβαστική 5 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά να ελέγξουμε λοιπόν ψηφίζουμε τη συμβαστική 5 πέρασε Όχι, απορρίπτεται. Α, δεν λειτουργεί κάποιο μηχάνημα. Αλλά όπως και αν ψηφίσατε είναι 20 ε, κατά και 18 υπέρ. Και επιπλέον είστε κατά κι εσείς. Λοιπόν, απορρίπτεται η συμβαστική 5. Πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία τις τροπολογίες που κάλυπτε. Λοιπόν, λοιπόν ξεκινάμε. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ελέγχουμε την 305 άρχεται πέρας εγκρίνεται 304 304, 33 και 36. Αυτές καταπίπτουν λοιπόν. Πάμε στην 306. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 306. Πέρας. Απολύπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές άρχεται η ψηφοφορία για την 34 πέρας απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά Άποχες. Δεν είναι σαφές και πάλι ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η 1. 303. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι καθόλου σαφές. Μα τι, μα τι λέει κύριε Βαντεκά, πώς είναι σαφές. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την συμβαστική 5α. Πέρας. Υπάρχει πολύ ευρία πλειοψηφία. Είτε είστε λίγο κουρασμένοι και δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Ήδη κύριε Βαντεκάμπ, ήδη. Εγκρίνεται λοιπόν έλεγα. Λοιπόν συνεχίζουμε. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τριάντα εννέα. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε. Ελέγχουμε την 39. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε μαζί τις 19, 37, 72, 73, 74, 75 και 76. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεν εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ε, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20-20. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 3.17. Υπέρ παρακαλώ. Κατά άποχες. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ε, ούτως άλλως θα, θα μου ζητήσετε έλεγχο, οπότε εγώ ξέρω ότι έχει απορριφθεί, αλλά ο κύριος Ρικέ μου ζητάει ε, έλεγχο και επειδή είμαι δημοκράτης ε, να ελέγξουμε την 317. Πέρας. 20-20. Μα το είχα πει. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 8. Κατά αποχές Ποιος είπε δεν είναι σαφές. Κύριε Καλάρε, εσείς το είπατε. Ωραία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Για τη συμβαστική 8. Πέρασε. εγκρινεται Εγκρίνεται. 22-17. Λοιπόν, 3.42 υπέρ κατά άποχες Λοιπόν, ελέγχουμε Πέρας Εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές άρχεται πέρας εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 362 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 10α υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τετρακόσια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.13 υπέρ κατά άποχες ασαφές ελέγχουμε την 4.13 πέρας εγκρίνεται 53 υπέρ κατά άποχες Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 53 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 4, 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 57 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 444 υπέρ. 444. Αγιάλα, κυρία Αγιάλα Σέντερ. Αμέσως μετά τη συμβαστική 12. Εντάξει κυρία Αγιάλα, άριστα. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλά, λοιπόν, ελέγχουμε. Την 58. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 468 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 466 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε την 466 άρχεται πέρας Α, απορρίπτεται. Λοιπόν, περνάμε στα παραρτήματα. 4,70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε κατευθείαν στην 480 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές. Ελέγχουμε την 480. Πέρας. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο της 63. Καλώς. Άρχεται. Πέρας. όπως είχα πει εγκρίνεται. Να με εμπιστεύεστε. Λοιπόν, 77 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Κύριε Βαντεκάμπ, καλά, καλά, ελέγχουμε, άρχεται. Την 80. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν με πιστεύεστε κύριε Βαντεκάμπ. Όχι δημοσίως όμως. Τουλάχιστον να είστε διακριτικός. 81. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά άποχες νομίζω απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε την 82 Πέρας. 20 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία MV2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. MV4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. NV5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τις 2 και 3 από κοινού υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνονται. Οπότε πάμε στην ένβη 7, όχι 10, 10. Ένβη 10 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι δύο της κυρία Γιάλα Σέντερ 103 και 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 104 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, 104 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές ασαφές ελέγχουμε την 113 πέρας απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω οπότε ελέγχουμε την 116 πέρας απορρίπτεται με ισοψηφία 20 8 υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ελέγχουμε την οκτω Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ένα, 1-1-4 υπέρ. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Συγγνώμη κυρία Ταπαρτέλ, δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία σας. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Πάλι εσείς κύριε Βαντεκάμπ. Καλά. Ελέγχουμε. Την 10. Πέρας. Κύριε Βιν Βαντεκάμπ, εγκρίνεται. Δεκατέσσερα 14-16 14. Ψηφίζουμε την 16 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 όμως καταπίπτει. Η 12 υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, παρακαλώ, λίγο περισσότερη συγκέντρωση. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές με συγχωρείτε ε, λίγο πιο σιγά παρακαλώ γιατί ψηφίζουμε ευχαριστώ πολύ λοιπόν ξεκινάμε πάλι 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλά ελέγχουμε την 173. Πέρας. Ισοψηφία. Καλά που είστε εδώ κύριε Κορ. Απορρίπτεται. 174. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 ταυτόσημες 186 και 187 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται συμβαστική 23 υπέρ 23 λέω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται να ψηφίσουμε το κείμενο συνολικά και ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρασε. Υπέρ 35, κατά 2 και 3 αποχές. Συγχαίρουμε την κυρία Γονταλόν. Εγκρίνεται η έκθεσή σας. Κυρία Ριβονταλόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να σας ζητήσω μια πολύ μικρή διακοπή για λίγα λεπτά. Πρέπει να συνεννοηθώ πολύ γρήγορα με τους κοιόδης. Πρόεδρος. Ωραία λοιπόν. Θα ζητήσω από τους εισηγητές και τους συνεισηγητές να βγουν για λίγο από την αίθουσα επειδή πρέπει να συνεννοηθούν και θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για αυτό το λόγο. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την, ε, ψηφοφορία μα, μας, παρακαλώ. Κύριε Βαντενκάμπ, ήδη... Ε, κυρία Ριβόντα Λόν, ε, μετά από συνεννόηση με τους διάφορους σκιώδεις εισηγητές, ήθελα να σας προτείνω να ψηφίσουμε και την εντολή για την έναρξη προμοτεύσεων. Εντάξει λοιπόν, ως πρόεδρος δέχομαι το έτοιμά σας, οπότε να ψηφίσουμε την εντολή για να περάσετε σε τριμερή διάλογο. Ε, ανοίγει η ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται αυτή. Χρειαζόμαστε 25 ψηφίσαντες, πέρας. Έχετε πάνω από 38 ψήφους υπέρ. Εγκρίθηκε η εντολή. Πάτε απευθεία στον τριμερή διάλογο. Μπράβο σας κυρία Ριβονταλόνη. Να συνεχίσουμε. Έκθεση κλούν. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομή όσον αφορά ορισμένε διατάξει σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων. Κυρία Κλούν, καλημέρα σα. Καλά είστε. Είστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Δεν ψηφίζουμε την τροπολογία 10, η οποία καταπίπτει. Τροπολογία της Επιτροπής ΑΕΚΟΝ 2, προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Όχι. <coughs> Οπότε ψηφίζουμε την προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί 4, 5, 32, 4, 6, 34, 5 της Επιτροπής ΕΚΟΝ, 7, 36, 6, 8, 38, 7, 9, 41, 8, 3. Δεν αποφασίζεται ε, εάν είναι αναγκαίο ή όχι. Εγώ θα ήθελα να είμαι βέβαιη ότι η αριθμη είναι σωστη σε όλου του καταλόγου προφοριών. Ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Δεύτερο μπλοκ. 33-37. Όχι. Καταπίπτει. Διότι μόλις εγκρίναμε το προηγούμενο. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 δεν ψηφίζεται. 27 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 απευθείας. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 32 υπέρ, 4 κατά, 2 εποχές. Μπράβο σας κυρία Κλούν, εγκρίθηκε η έκθεσή σας. Συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Σαλίνη πρόταση οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση. Κύριε Σαλίνη, είστε έτοιμο. Πάμε. Συμβαστική πρώτη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση. Κύριε Ρικέ. Για την Λίμπε 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίμπε 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. 31 υπέρ. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Εγκρίνατε. Με συγχωρείτε. Όχι 71. Προέτρεξα. 68. Και 69 και 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Δεν με σήμερα. Ωραία λοιπόν να ψηφίσουμε τις τρεις τροπολογίες αυτές. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. 27 κατά. Απορρίπτονται. Να συνεχίσουμε. 71. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ 73 υπέρ Δεν είστε υπέρ της απολογίας σας κύριε Βαντεκάμπ. Εντυπωσιακό. κατά της τροπολογίας Βαντενκάμπ. Πλειοψηφία απορρίπτεται. Συνεχίζουμε 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ταυτόσιμες οι εξής δύο. 76-77 υπέρ κατά αποχές κρίνονται. 78. Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απευθείας περνάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 απευθείας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απευθείας τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. Επαλήθευση για την 108. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 ταυτόσημες 112 και 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Εκατόν δεκαεννέα, υπέρ. Κατά. Είστε κουρασμένοι μου φαίνεται. Για να ξαναρχίσουμε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 α καταπίπτει 120 απευθείας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι κάνετε κύριε Ρικέ. 121. Δεν φάνηκε. Ε, ξαναψηφίζουμε. 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Απευθείας 126 τώρα. Υπέρ. Κατά. Είστε λίγο χαμένοι μέσα στα χαρτιά σας. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4α, συμβαστικά 4α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απευθείας 140 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές 141 δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει Άρια την ψηφοφορία ηλεκτρονικός πέρας εγκρίνεται Λίμπε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Να ελέγξουμε 21 για Λίμπε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγ... απορρίπτεται. 22 λίμπ 22 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Λίμπ 22. Πέρας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 146 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται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 αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας 20-20 22-20 Είχα δίκιο, εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. Απευθεία, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 27 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός λίμπε 27 πέρας απορρίπτεται Τροπολογία 13 και 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Απευθείας. Λίμπε 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες 166-167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Λίμπε 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με τη λογική σκέψη. Λίμπε 1 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση λίμπε 1 πέρας 21-21 ισοψηφία απορρίπτεται. Λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 56 καταπίπτει, 54 απευθείας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας. 40 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σαλίνη. Et nous votons dans la foulée le mandat και ψηφίζουμε μαζί και την εντολή, τη δημοτευτική εντολή. Θα χρειαστεί πλειοψηφία 25 ε, ψήφων. Ψηφίζουμε την εντολή λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Je ferme le vote. Πέρας. η πλειοψηφία είναι και περισσότερο από απόλυτη. 41 υπέρ, ε, έχετε απόλυτη ελευθερία για να πάτε για διαπραγματεύσει. Τώρα το φορτίο είναι στους δικούς σα όμω, κύριε Σαλήνη. 41 συνάδελφοι υπέρ, όλοι συμφωνούν για να περάσετε σε τριμερεί διαλόγους και σα στηρίζουν. Ευχαριστώ Ντομινίκ. Και τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση της κυρίας Μοντέιρο. Έκθεση Μοντέρο αφορά την χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Καλημέρα σας κυρία Μοντέρο, είσαστε καλά. Προχωρούμε, ξεκινούμε. Ένα α, υπέρ. Le compromis 1A. Ξανά πάλι, ένα α, υπέρ. Contre. Qui s'abstient. c'est pas clair. Όχι, δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα, οπότε θα γίνει ηλεκτρονικό έλεγχο για τη συμβαστική 1α. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και προχωρούμε στη συμβαστική 2α υπέρ. 2α. Υπέρ, κατά, α, αποχές. ίδια πλειοψηφία νομίζω. Αλλά ζητείτε την επανλήθευση. Ναι, ναι, βεβαίω, βεβαίω. Ψηφίζομαι. Πέρασε. ίδια πλειοψηφία.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 Δεν πρόκειται για πάρτι. 3α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, οπότε θα κάνουμε έλεγχο για το 3α. Πέρασε ο ψηφοφορίας. Συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Το 3α επόμενο συγκεντρώσει. Και τώρα προχωρούμε στο 74 υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ του 74. Τροπολογία 74. Να mais mettez-vous d'accord, on recommence. Βρείτε τα, βρείτε τα. Και πάλι. Εκεί η παρέα, ναι, να, να το γλεντάτε, αλλά να είστε συγκεντρωμένοι υπέρ του 74, κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική 74. Ψηφίζουμε. Je ferme le vote. Απορρίπτεται. Παρακάτω. Συμβαστική 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 72 υπέρ κατά αποχές δεν σαφές το αποτέλεσμα επαλήθευση για το 72 πέρας απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο των τροπολογιών όσον αφορά το 38, 39, 61, 71, 73, 75. Υπέρ. Κατά αφορούν τους τίτλους αυτές οι τροπολογίες. Επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτονται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ζητείτε ηλεκτρονικός έλεγχος. Madame Anderson. Κυρία Άντερσον, προσέξτε το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Allez, nous allons vérifier, parce que là... Αν να κάνουμε επαλήθευση, τότε ψηφίζουμε για το 79. Oui, oui. Je ferme le vote. Πέρασε ο Απορρίπτεται. 80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 Mais vous êtes rieur aujourd'hui, hein Allez, on continue. Amendement 14. 14, υπέρ. Συμπαθάτε με γιατί έκανε κάποιο λάθο λέει ο Πρόεδρος, γιατί ψηφίσαμε το 80 και περιευθεί, αλλά δεν ψηφίσαμε το 81. Οπότε το ψηφίζουμε. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει επαλήθευση. 81. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. 32. Qui est pour Attendez, attendez, attendez. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Όχι καταπίπτει. Άρα το 32 δεν το ψηφίζουμε, πάμε 34 υπέρ. Qui est qui s'abstient. κατά εγκρίνεται και τώρα το σύνολο της ε, έκθεσης. Ψηφίζουμε. Πέρας. 24 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίθηκε η εκθέσή σας κύριε Μοντέιρο. Και τώρα θα ψηφίσουμε την διαπραγματευτική εντολή. Le mandat de négociation Είναι για τον τριμερή διάλογο. Κύριε Μοντέρο, θέλετε και το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απλώς να ζητήσω και εγώ για δύο λεπτά να διακόψουμε και να συνεννοηθούμε με τους ε, σκιώδεις. Για την ε, εντολή, λέει Πρόεδρος, περιμένετε γιατί κάνουμε μια μικρή διακοπή πεντάλεπτη. discutez, vous discutez dehors. Οι κουβεντούλε έξω. La parole est à vous. Έχετε το λόγο, κυρία Μοντέιρο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να περάσουμε στην πληροφορία για την δημοκρατική εντολή. D'accord. Πολύ ωραία λοιπόν και τώρα θα θέτουμε η ψηφοφορία την διαπραγματευτική εντολή για την έκθεση Μοντέιρο.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 Mes chers collègues, nous allons reprendre... Κύριε Πρόεδρο, συνεχίζουμε τις εργασίες μας, συνάδελφοι. Allez, nous commençons. Αρχίζουμε. Κύριε Βαντεκάμπ. Allez, nous commençons avec la proposition de directive. Έχουμε το σχέδιο οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία του 2009, υπαριθμών 33, για οχήματα οδικών μεταφορών καθαρών και αποδοτικών ενεργειακά. Ο εισηγητής έχει το λόγο, ο κύριος Αντόρ Ντέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, very that φανερό έχει καταστεί ότι η οδηγία 29 κάθετος 2009 κάθετος 33 ε, θα έπρεπε να τροποποιηθεί και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ευτυχώ που έφτασε η πρόταση Ευρωπιστοτικής γιατί λόγω της εκ των υστέρων αξιολόγησης που έγινε το 2015 ξεκάθαρα πρόκειπτε ότι ιστερούσε η ρύθμιση και ο σκοπός της ε, τροποποίησης ήταν σημαντικός διότι το πνεύμα που διέπνε την πρόταση της Επιτροπής ήταν το να δώσει μια όθηση στην αγορά καθαρών και χαμηλών εκπομπών οχημάτων μέσω του κρατικού τομέα, γιατί έτσι θεωρήθηκε ότι θα αναπτυχθούν υποδομές και έτσι θα τονωθεί η αγορά γενικότερα. Όταν συνέταξα την γνωμοδότηση, συνέταξα και 26 τροπολογίες. Επί της ε, ουσίας αυτών των τροπολογιών Οφείλω να σας πω ότι αυτό που ήθελα ήταν να διευρύνω το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τα οχήματα τα οποία θα εκαλύπτονται από την προ... Οπότε έτσι ε, κάλυψα και τα ταξί, τα οχήματα, ε, τα ελαφρά φορτηγά, ε, επίσης τα μισθωμένα οχήματα γιατί θεώρησα ότι το ότι ήταν αρκετά στενό το πεδίο εφαρμογή αποτελούσε από τα προβλήματα της ε, οδηγίας οπότε με την ε, τροποποίηση θα έπρεπε να επιφέρουμε αυτή την μεταβολή τώρα όσον αφορά κάποιες ε, παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις ήδη η Κομισιόν είχε κάποιες τεκμηριωμένες τέτοιες εξαιρέσεις αλλά εγώ πρόσθεσα και άλλες γιατί προέκυψε σαφώ ότι υπήρχαν κάποια μισθωμένα από το δημόσιο οχήματα τα οποία θα έπρεπε να εξαιρεθούν και μιλούμε για κάποια οχήματα τα οποία είναι ειδικών σκοπών και έχουν ειδικό σχεδιασμό αποχετεύσεις, νερό, ε, συντήρηση ηλεκτρολογικού δικτύου, ε, ασφάλεια, ε, κατεπίγουσες καταστάσεις όπως πλημμύρες, ε, πού να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες περιπτώσει πλημμυρών τα ηλεκτρικά οχήματα. Πρώτα πρόσθεσε αυτές τις εξαιρέσεις στην πρόταση της Επιτροπής υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις με την οδηγία για εναλλακτικά καύσιμα. Άρα συνεκρούντο η οδηγία εκείνη με την παρούσα και αυτό αφορά τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και για αυτό το λόγο και πρότεινα έναν ορισμό ο οποίος θα μπορούσε να συνάδει με την οδηγία εκείνη για τα εναλλακτικά καύσιμα και τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών σε σχέση με αυτά τα επιλέξιμα καύσιμα επίσης. Σε σχέση με τους ε, επισυναπτώμενους πίνακες για τα εθνικά κατόφλια όπως ε, διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ έθεσα κάποιους ε, στόχους ελαχίστων εκπομπών, ελαχίστων οριακών τιμών τέλο πάντων για την κοινότητα σε σχέση με τα παλιά και τα νέα κρατημέλη γιατί είχαμε ε, κάποια κατόφλια τα οποία ακριβώ απήχαν για τις μεν χώρες από τις δε είπαμε ότι αυτά τα ελαφρά οχήματα L και λοιπά είπαμε ότι θα πάμε στο 25% με όριο το 2025 ούτω ώστε να καλύψουμε τις χαμηλές και τις μηδενικές εκπομπές. Πάντως η τιμή στόχος για 25 έως 30 θα μείνει ο ίδιο 25% αλλά να καλύψουμε μόνο τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και όχι τα οχήματα χαμηλών εκπομπών. Επίσης, σαφώς προέκυπτε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την μέθοδο υπολογισμού ήταν μάλλον περίπλοκη. Οπότε, είπαμε να αποφευθεί η περαιτέρω σύγχυση και πρότεινα το εξής τουλάχιστον το 2025 όλα τα οχήματα να μετρούν ως ένα. Και το χειμώνα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Και στη συνέχεια ως ένα όχημα να είναι μόνο τα μηδενική ε, εκπομπής οχήματα. Τώρα όσον αφορά τα, βα, τα οχήματα, τα, τα βαρέα φορτηγά εδώ θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ λεωφορείων και φορτηγών γιατί όσον αφορά τα φορτηγά δεν έχουμε τη σχετική αγορά, δηλαδή φορτηγά με μηδενικές συμβόντες. Όμως, στα ε, στα λεωφορεία, άλλα ισχύουν. Έχει εξελιχθεί περισσότερη κατάσταση, άρα θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των μεν και των δε οχημάτων και επομένω ε, θα πρέπει η τιμή στόχος να μείνει στο 10% για τις προμήθειες και έτσι να καλύψουμε και τα ε, οχήματα αυτά αλλά το 10% να γίνει 15% μέχρι το 2030. Στον αυτά τα φορτηγά για τα λεωφορεία τώρα μέχρι το 2025 να είναι 35% για κάθε προμήθεια και μέχρι το 2030 θα πρέπει να πάμε στο 70% για τα λεωφορεία χαμηλών και μηδενών εκπομπών. Τώρα, όσον αφορά τις αιτιολογικές παραγράφους 2, την έχω να σας πω, ήταν σαφές ότι η οδηγία αυτή είχε σχέση με τις μετρήσεις εκπομπών για διοξίδιο, για άζωτο, με τη συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης, αλλά εγώ ήθελα να αλλάξουμε προσέγγιση και θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και άλλα στοιχεία. Πάντως αυτό τώρα δεν είναι στο σώμα της οδηγίας, αλλά στην ιδεολογική παράγραφο. Και έτσι να δείξουμε στην Κομισιόν τι δρόμο θέλουμε να πάρει πρότασή της. Κάτι άλλο τώρα. Και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη σε διάφορα επίπεδα θα πρέπει να δώσουν περισσότερα κίνητρα και δεν μιλώ μόνο για τα οικονομικά κίνητρα αλλά τα κίνητρα γενικότερα αυτά λέω σε αιτιολογική παράγραφο και ελπίζω ότι με τις προπολογίες αυτές μπορούμε να έχουμε τεχνολογικά ουδέτερη πρόταση. Γιατί μπορούμε να έχουμε μηδενικές εκπομπές και από άλλα καύσιμα, όχι μόνο με ηλεκτρισμό. Υδρογόνο, ε, καύσιμα που δεν είναι ορυκτά, Έχουμε, έχουμε επιλογές διάφορες. Και έχουμε έρευνες που χρηματοδοτεί η Ένωση. Άρα δεν θα πρέπει να πηγαίνουν χαμένα όλα αυτά τα χρήματα. Περιμένω πώς και πώς συναδελφοί τη γνώμη σας, αλλά περιμένω και τις τροπολογίες σας που θα ακολουθήσουν. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Άντερσον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις αναλυτικές εξηγήσει τη έκθεση του που μόλι μα έδωσε. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν. Πολύ σημαντικό μέτρο. Και προσβλέπουμε στην ε, συνεργασία με τον εισηγητή για να υπάρξουν αλλαγέ. Οι δημόσιε προμήθειε είναι πολύ σημαντικό. Δεν καλύπτει όλο τον ιδιωτικό τομέα βεβαίω, αλλά έχουμε πολλά στοιχεία παντού στον κόσμο ότι οι δημόσιες προμήθειες παίζουν σημαντικό ρόλο γενικά για να έχουμε πιο καθαρά οχήματα αλλά και σε άλλους τομείς. Και από ό,τι ακούμε από τους κατασκευαστές έχουν πρόβλημα γιατί συχνά δεν έχουν τα αυτοκίνητα που θα ήθελαν να κατασκευάσουν. Η έκθεση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή οδηγία. Να γίνει όσο ευρύ γίνεται λογικά. Και γενικά νομίζω ότι οι κατηγορίες οχημάτων που συμπεριλαμβάνονται όπως και τα ταξί είναι πολύ ε, σωστές. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τι εξαιρέσεις θα δώσουμε. Δεν είναι μόνο ε, η διεύρυνση, αλλά πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε οι εξαιρέσεις να μην έχουν αθέλητες αρνητικές επιπτώσεις. Και επίσης πρέπει να δούμε και τις εκπομπές ε, στα εργοτάξια στις πόλεις, που είναι πρόβλημα σε πολλές πόλεις, όπως τη δική μου. Πρέπει να το δούμε. Και με, το, με τα διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις ε, κατασκευές. Καταλαβαίνω το στόχο απλούστευσης τώρα, τώρα για κάποιους ορισμούς, αλλά δεν συμφωνούμε, τουλάχιστον ε, σε μια πρώτη φάση, με την απλούστευση που θα το προσαρμόσει στις τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να καταλήξουμε ε, σε κάτι το οποίο θα γίνεται παροχημένο πολύ σύντομα. Ε, πρέπει φυσικά να είναι τεχνολογικά ουδέτερη η προσέγγιση μας. Για τους στόχους τώρα συγκεκριμένα πρέπει να είμαστε όσο πιο φιλόδοξοι γίνεται. Και για να είμαστε φιλόδοξοι θα πρέπει να δούμε και τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Mm και να έχουμε διαφοροποιημένους λοιπόν στόχους, ανά κράτος, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν σε ενωσιακό επίπεδο τις δυνατότητες. Πρέπει επίσης να υπάρχει και αυτή η ρήτρα αναθεώρησης και να είναι πιο κατηγορηματική. Να μην ε, καθυστερούμε αυτές τις αναθεωρήσεις, γιατί αυτό είναι πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Αν το Κοινοβούλιο έχει πιο ρωμαλαία προσέγγιση, για τις αναθεωρήσεις νομίζω ότι θα βοηθήσει την Επιτροπή. Και πολλά άλλα σημεία, απλώς δειγματοληπτικά ανέφερα ορισμένα, αλλά θα τα συζητήσουμε πιστεύω και θα καταλήξουμε πολύ θετικά. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Ο κύριος ε, Ντόλσον. Έχει, έχει το λόγο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Και εμείς ε, καλωσορίζουμε αυτήν την ε, μεταρρύθμιση. Όπως είπε ο συγητής, ε, η υπάρχουσα οδηγία είχε πολύ λίγη εφαρμογή, πολύ μικρή εφαρμογή. Μέσω της αναθεώρησης μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους της αρχικής νομοθεσίας. Όμως οι αρχικές προτάσεις ε, δεν περιλαμβάνουν σωστούς ορισμούς και θέτουν ε, στόχους για τις δημόσιες προμήθειες που δεν λαμβάνουν υπόψη την εξελισσόμενη τεχνολογία. Η πρόταση βεβαίως διευρύνει το φάσμα και καθορίζει τα καθαρά οχήματα σύμφωνα με τις ε, ρήτρες της ε, οδηγίας Ντάφη. Τον στηρίζουμε λοιπόν για την εργασία του μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα, ώστε να είναι και αποτελεσματικές και σωστά ε, προσαρμοσμένες με την πραγματικότητα οι προτάσεις. Ιδιαίτερα λοιπόν πρέπει να δούμε τους στόχους. Πρέπει να δούμε πώς αναπτύσσεται η αγορά για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Είναι πολύ ακριβά αυτά τα οχήματα τώρα. Υπάρχει πολύ περιθώριο για τεχνολογική πρόοδο, ούτω ώστε να προσαρμοστούν αυτοί οι στόχοι για τις δημόσιες προμήθειες στην πραγματικότητα της αγοράς. Υπάρχει ένα παράδειγμα που ξέρει και η Λούση πολύ καλά. Τα καινούργια ταξί στο Λονδίνο. Οι οδηγοί μπορούν να αγοράσουν τώρα μόνο ηλεκτρικά ταξί. Είναι πολύ καλά ταξί. Φτιάχνονται στην εκλογική μου περιφέρεια, πολύ καλά, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά και πολλοί ταξιτζίδες στο Λονδίνο δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Άρα δεν θα τα αγοράσουν και θα συνεχίσουν να εκλοφορούν τα παλιά ταξί. Αυτό τελικά ε, είναι αντιπαραγωγικό. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε αρκετά κίνητρα ε, για να πάρουν καινούργια οχήματα, ε, ιδίω οι ταξιτζίδε, αλλά και για καινούργια λεωφορεία, γιατί οι πόλει με προβλήματα προπολογισμού δεν θα μπορούν να τα αγοράσουν. Δεύτερον, οι ορισμοί σε όλο το πακέτο καθαρής κινητικότητας θα πρέπει να, είναι, να συνάδουν με την οδηγία DAFI. Ε, και βεβαίω πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ουδετερότητα. Βεβαίω τα ηλεκτρικά οχήματα θα παίξουν τεράστιο ρόλο και όλοι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τα ηλεκτρικά οχήματα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τα βιοκαύσιμα δεύτερη δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τα βιοκαύσιμα γενιάς και άλλες ε, ε, άλλοι κινητήρες εσωτερικής καύσης, ιδιαίτερα του ντίζελ, γίνονται όλο και πιο ε, καθαροί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τους συμπεριλάβουμε και αυτού γενικά. Στηρίζω όμως ε, την έκθεση Ντάλι και προβλέπω στη συνεργασία μας και τους κοιόδης βεβαίω, γιατί πιστεύω ότι θα επιτύχουμε πολύ θετικέ συμβαστικές τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τελίτσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Να πω ότι γενικώ η προσέγγιση του συγητή με καθησυχάζει, παρόλο που θα ήθελα σε κάποιες από τις λεπτομέρειες να υπάρξουν διευκρινήσεις. Η πρώτη μου παρατήρηση απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συμφωνώ με την αναθεώρηση τη οδηγία του 2009, αλλά νομίζω ότι μακροπρόθεσμα ως αντιδρα... Ε, ε, η σωστή αντίδραση θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει έμφαση στα στοιχεία όπου θα πρέπει να δούμε πού ε, δεν υπήρξε καλό αποτέλεσμα γιατί υπήρξαν σημεία συμφόρησης για να έχουμε τις απαραίτητες ε, κατευθυντήριες γραμμές. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η τεχνολογική οδετερότητα. Τίνουμε να λέμε μηδενικές εκπομπές και το συνδέουμε αυτό με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Όμως δεν είναι εντελώ ε, απαλλαγμένα από εκπομπές τα ηλεκτροκίνητα. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν συνολικά την εικόνα του περιβάλλοντος στην Ένωση, και δούμε και την προοπτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Είναι υπερβολική και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή κυρίω επικεντρωνόμαστε στα ηλεκτροκίνητα και αυτό φαίνεται και ο ρόλο αυτή τη αναθεώρηση. Εγώ όμω νομίζω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο να πετύχουμε αποτελέσματα στα δυνατό συντομότερα. Δηλαδή να ασχοληθούμε με το στόλο όλων των οχημάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εάν ε, θα επιλέξουμε τα ηλεκτροκίνητα πάνω από όλα ή τις μηδενικές εκπομπές είναι άλλο θέμα, αλλά πρέπει να δούμε και τη μέση ηλικία των οχημάτων και το μέσο όχημα που βρίσκεται στην αγορά. Αυτό είναι ένας λόγος ακόμα που η τεχνολογική ουδετερότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα σε μια συνολική εικόνα και σε σύγκριση με το τι ήδη υπάρχει στην αγορά. Για μένα αυτό είναι ζωτική σημασία. Και θα πρέπει να σταθούμε με προσοχή στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή ήταν η δεύτερη παρατήρηση. Τώρα, ως προς τους στόχους αναχώρα, έχω κάποια συμπάθεια για την προσέγγιση του εισηγητή, όμως η Επιτροπή θα μπορούσε ίσως να διευκολύνει τα πράγματα. Δεν με ενοχλεί να τα λέτε μεταξύ σα, αλλά είναι κάπως ενοχλητικό, εάν μπορείτε να με προσέχατε λίγο. Τα κριτήρια που έχει χρησιμοποιήσει ο, η Επιτροπή για το στόχο αναχώρα. βεβαίω το ΑΕΠ είναι βασικό, το βασικό κριτήριο. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν τελείω διαφορετική νομοθετική διοργάνωση τα διάφορα κράτη-μέλη και βάσει του συνταγματός του. Αυτό θα πρέπει να το δει προσεκτικά η Επιτροπή. Έχει ληφθεί υπόψη γιατί έχει ένα επιχείρημα ο εισηγητή, έχει προβάλλει ένα επιχείρημα όπου μιλάει για ενδεχόμενη απαλληφή των ε, στόχων αναχώρα. Επίσης το σχέδιο της έκθεσης κάνει λόγο για κίνητρα. Θα προσπαθήσω να το αναπτύξω, αλλά μήπως πρέπει να σκεφτούμε έναν ενδεικτικό κατάλογο ε, κινήτρων που θα μπορούσαμε να προτείνουμε δηλαδή ένα παράρτημα, ε, ενό είδου παράρτημα που εφόσον προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρα αυτά που θα προτείνουμε. Τώρα για τις κατηγορίες των οχημάτων συμφωνώ με τη βασική προσέγγιση. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά τις κατηγορίες πιο ευρέως, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στις εξαιρέσεις που θα προτείνουμε για την δίτροχη προσέγγιση ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες σε αυτήν την αναθεώρηση. Η δυσκολία, η συμφόρηση ε, που θα προκύψει από ε, την συνάντηση πολλών διαφορετικών στοιχείων είναι οι υποδομές. Θα κοιτάξω αν μπορώ να δώσω έμφαση σε αυτό το θέμα και να ε, υποβάλω σχετικά τροπολογίες για τις λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ ολοκληρωμένο κείμενο με τη συμβολή όλων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Τέλετσκα. Είχα εγγραφεί και εγώ στον κατάλογο των αγορητών γιατί δεν είναι εδώ ο κύριο Νταλούντε και ζητά συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Ντέλε για την έκθεσή σα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια αλλαγή του μοντέλου της νοοτροπίας ε, που επικρατεί για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα αυτοκίνητα του παρελθόντος δεν μπορούν πια να παράγονται. Η έκθεση λοιπόν αυτή ε, αναπτύσσει και μια θεώρηση για το μέλλον. Με ένα στόχο, ε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα, από την ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Είναι ένας πολύ χειροπιαστός στόχος. Εάν σε αυτήν την επιτροπή καταλάβουμε ε, και υποδεχτούμε ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα ορεικτά καύσιμα, θα πρέπει κάπως να προλάβουμε από τώρα. Και κάποιες φορές έχουν εντύπωση ότι δεν θέλουμε να προλάβουμε, διότι κάποιοι λένε ότι υπάρχει το βιοντίζελ ή τα βιοκαύσιμα. Στα βιοκαύσιμα και στο βιοντίζελ το μόνο βιολογικό στοιχείο που έχουν, το μόνο οικολογικό είναι το όνομά του. τίποτα άλλο. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Γιατί, Γιατί πάρει κανεί το βιοντίζελ, α πούμε, η βάση σύνθεση του ε, βιοντίζελ είναι το φινικέλαιο. Το φινικέλαιο ε, απαγορεύτηκε από αυτό το κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να το απαγορεύσει εντελώ από το 2021. Δεν θα μπορούμε πλέον να ακολουθούμε τέτοιες ε, άγουσες διότι θυμίζω ότι το Φινικέλ είναι τρεις φορές ε, πιο επιζήμιο για το κλίμα και καταστρέφει εκτάρια τροπικών δασών επί εκταρίων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, υπαναχωρήσουμε σε σχέση με αυτή την απόφασή μας. Ως προς τους οικονομολόγους όλοι λένε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Στην, έκθεση αυτή, στην Επιτροπή αυτή είχαμε μία ε, έκθεση σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια και τα ηλεκτροκίνητα που δείχνει ότι δεν είναι τόσο οικονομικά τα οχήματα αυτά. Τα ηλεκτροκίνητα από μόνα τους δεν θα είναι η μόνη λύση για να ξεφύγουμε από όλα τα προβλήματα ρήπανσης και ούτω καθεξής. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να επινοήσουμε ένα νέο ενεργειακό μίξ. Όταν μιλάμε για υδρογόνο, ας πούμε, για αέριο, φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι ιδέες για το μέλλον. Τρίτο στοιχείο που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι τα οικολογικά αυτοκίνητα του μέλλοντος θα είναι ε, οικολογικά αν είναι από το α ως το ω ανακυκλώσιμο. Το πρόβλημά μας σήμερα είναι ότι κανένα κομμάτι της κυκλικής οικονομίας δεν έχει αξιοποιηθεί για να ανακυκλωθούν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα. Επίσης ένα ε, όχημα οικολογικό στο μέλλον θα είναι ένα όχημα που δεν θα είναι γιοταχή. Θα είναι ένα όχημα ε, μοιρασμένο μεταξύ περισσότερων χρηστών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και ένα σύστημα για την ε, κοινοχτημοσύνη κατά κάποιο τρόπο των οχημάτων. Επίση έχουμε 13 εκατομμύρια ε, χρήστες στην Ευρώπη, ε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να πέραν από τι λύσει που θα προτείνουμε να προβλέψουμε και την εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι οικολογικέ μα λύσει θα πρέπει να υποστηρίζονται από τι τεχνολογικέ εξελίξει, νέε τεχνολογίε. Αυτό απαιτεί εκπαίδευση, απαιτεί γνώσει που σήμερα δεν είναι απαραίτητα δεδομένε για όλου του εργαζόμενου. Και Τρίτο, και που για μένα είναι το πιο σημαντικό, τι θα κάνουμε με τα οχήματα που σήμερα κυκλοφορούν, που δεν σέβονται τους κανόνες Euro 6. Αυτό είναι ένα κατεπήγον πρόβλημα και αυτή είναι μια βόμβα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη. Το είδαμε με τον Dieselgate, το σκάνδαλο του, της Volkswagen. Ε, πολλά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους μας σήμερα είναι πραγματικά για τα σκουπίδια και ξεπερνούν τα όρια όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές, αλλά 17 φορές. Ε, τι κάνουμε λοιπόν με αυτά τα εκατομμύρια αυτοκίνητα. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι η έκθεση αυτή όταν λέμε εξοικονομούν ενέργεια οικολογικά και το καθεξής πρέπει να προτείνει και μια λύση για τα σημερινά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους σήμερα. Για να ε, μη βρεθούν ε, σε ε, χώρους αποκομιδής ε, κάπου μακριά στην Αφρική όπως καταγγέλει ο τύπος ε, και είναι αυτό η λύση που προτείνουμε. Ένα κύκλο των αυτοκινήτων αυτών σημαίνει ότι τα σημερινά ε, οχήματα σήμερα θα έπρεπε να μπορούν να μετατραπούν αύριο σε ηλεκτροκίνητα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και ένα τέτοιο κλάδο παραγωγής να προτείνουμε. Εδώ κύριε Ντέλη, ε, οι δρόμοι που ανοίγουν η έκθεσή σας μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντες. Ελπίζω να πετύχουμε βήματα πρόοδου, αλλά να μην καταλήξουμε και σε αδιέξοδο σε κάποια σημεία όπου δεν καλύπτουμε παρκώς το θέμα. Κυρία Ντεπρέ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας δίνω ευθύ αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω καλωσορίζοντα την Επιτροπή σας για το έργο Είχαμε συνεννοήσεις και με άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Βλέπουμε ότι δραστηριοποιείται ιδιαίτερα το κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή. Είναι καλή ένδειξη. Και έχουμε καλές ενδείξεις για τη δουλειά που μας περιμένει και για την πρώτη ανάγνωση. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να ενισχύσουμε την καλή μας ως τώρα συνεργασία. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση του κυρίου Ντέλη να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία προς τους στόχους μας, την διεύρυνση του πεδίου σε σχέση με την τωρινή πρόταση. Ξέρουμε ότι θέλετε να πάτε πέρα από, από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι που το ανέφεραν και οι συναδελφοί σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και κάποια κάτι μέλη στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου που ασχολείται με το θέμα αυτό αλλά βλέπω ότι υπάρχει και στήριξη ως προς το να βρούμε ένα συγκεκριμένο ορισμό για τα καθαρά οχήματα, τα οικολογικά οχήματα, καθώς και τους στόχους για τους ελάχιστους όρους των δημόσιων προμηθειών. Σε ό,τι αφορά τους στόχους, ίσως υπάρχουν κάποιες μικροαποκλήσεις για τις διαφορετικές ομάδες, τέλος πάντων αυτά που προτείνουν οι σκιώδεις εξηγητές στην ουσία μεταξύ τους, αλλά υπάρχει από ό,τι φαίνεται η επιθυμία να διευρυνθεί το πεδίο σε σχέση με όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη όμως υπάρχουν ανησυχίες. Αυτό που λοιπόν θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι πρώτον είναι μια πρόταση που είναι τεχνολογικώς ουδέτερη. Προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες προμήθειες για να έχουμε ακόμα περισσότερη ή να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητα, εάν θέλετε. Επίσης, αυτά τα θέματα μας απασχολούν και στο Συμβούλιο και δεν ξέρουμε αν είναι καλή ιδέα να επαναχωρήσουμε στον ορισμό των εναλλακτικών καυσίμων από την προηγούμενη εκδοχή της οδηγίας. Το κοιτάζουμε. Αλλά εάν κοιτάξουμε τη διεύρυνση ε, του πεδίου σε αυτήν την οδηγία χωρίς πληρωματικά μέτρα θα χάσουμε από το επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Αυτό λοιπόν που συζητάμε στο Συμβούλιο είναι το κατά πόσον μπορούμε να επιδιώξουμε τις μηδενικές εκπομπές, τα οχήματα που θα έχουν μηδενικές εκπομπές, όχι τα ηλεκτροκίνητα, τα μηδενικών εκπομπών οχήματα. Και αυτό θέλω να το τονίσω εδώ, γιατί ο κύριος Ντέιλι το είπε. Έχουμε επενδύσει πολύ χρήμα για την έρευνα, για τις βιωσιμότερες τεχνολογικές λύσεις. Ε, πιστέψτε με, περιμένουμε ανυπόμονα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το υδρογόνο για τα μηδενικών κομπονοχήματα. Έχουμε δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα οχήματα. Ξέρετε ότι περιμένουμε αποτελέσματα από τις ερευνητικά μας κέντρα για να βγουν στους δρόμους. Οι στόχοι ανά μέλος, κάτι που ανέφεραν και η κυρία Άντερσον και ενώ πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ως προς το τι θέλουμε να πετύχουμε, ταυτόχρονα κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Και να απαντήσω και στον κύριο Τέλιτσκα. πώς καταλήγουμε στη φόρμουλα, στη συνταγή για να, διορίσουμε, να εντοπίσουμε διαφορές και απο, να καλύψουμε αποκλήσεις μεταξύ των 100 μελών. Εντοπίζουμε ένα ευρωπαϊκό μεσόωρο και μετά προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε τον στόχο Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με το ΕΠ και τον αριθμό του πληθυσμού. Διότι ο πληθυσμός είναι ένας τρόπος να δούμε πώς ε, διαμορφώνεται η ατμοσφαιρική ποιότητα και η ρήπανση σε διάφορες περιοχές. Ως προς την διεύρυνση του οχήματος και τις εξαιρέσεις Έχουμε κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να ξαναδούμε τις εξαιρέσεις. Στόχος, πάντως με τις εξαιρέσεις, δεν είναι να ρίξουμε το επίπεδο των φιλοδοξιών μας, απλώς να είναι η διάταξη σαφής, να είναι ξεκάθαρα το τι εννοούμε με το άρθρο αυτό. Και ίσως τελευταίο, α όχι, όχι, όχι, κάτι ξέχασα, για τον κύριο Τέλισκα. Ναι, γιατί η προηγούμενη οδηγία δεν ε, πέτυχε. Θα ήταν ε, επιπόλαιο να πούμε ότι οι αρχέ σε τοπικό επίπεδο δεν κοίταζαν παρά τι ελλείψει τη οδηγία πώ να αξιοποιήσουν τι δημόσιε προπήθειε για βιωσιμότερα οχήματα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι η ισχύουσα οδηγία δεν έχει πετύχει γιατί ίσως δεν υπήρχε και μια κοινή προσέγγιση για αυτά τα θέματα. Ως δημόσιες αρχές λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε ένα σαφές, μια σαφή ένδειξη στην αγορά, στις εταιρείε. Δεν τους προβάλαμε απαιτήσει, οπότε μείναμε λίγο στα ίδια. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Και αυτό ήθελα να το τονίσω. Και τελευταία παρατηρήση της κυρίας Μπελή για την ε, οικονομία επιμερισμού. Εδώ μιλάμε για δημόσιες προμήθειες οχημάτων, μισθώσεων, ε, αδειών που διαχειρίζονται δημόσιες αρχές. Έχω την αντιπόση ότι αυτό που αναφέρατε εσείς έχει να κάνει περισσότερο με το πώς περνάμε από το ΙΟΤΑΧΗ σε κοινή χρήση, κοινοκτημοσύνη ή τέλο πάντων ε, ταυτόχρονη αξιοποίηση των πόρων των μεταφορών. Αυτό έχει να κάνει με την ε, έκθεση πρωτοβουλία μου περισσότερο. Νομίζω ότι απήντησα στα περισσότερα σχόλια της αίθουσας. Ευχαριστούμε για αυτές τις παρατηρήσεις. Πριν σας δώσω το λόγο κύριε Τέλη, κύριε Τέλησκα, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Σας άκουγα απλώς εκεί που αναφέρατε την απορία σας για τα κριτήρια, ρωτούσα τον κύριο Ρικέ. Εάν δεν το είχαμε μόλις συζητήσει μεταξύ μας προηγουμένως και αν υπάρχει μέσα στην έκθεση ε, όχι. Το, το βρήκα πολύ ε, ε, ενδιαφέρον εγώ και περίεργο το να χρησιμοποιείται ως μόνο κριτήριο το ΑΕΠ. Σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη, αλλά σας παρακολουθούσα με προσοχή παρόλα αυτά. Κύριε Ντέλη. Uh, hear. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Με Διαβεβαιώσατε ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Για να σας πω την αλήθεια, ξέρω, ξέρω καλά ότι όπως σας τα είπατε η οδηγία αυτή έχει πολύ περιορισμένο βεληνικές. Πρόκειται για αυτές τις ε, προμήθειες από κρατικής πλευράς, τις νέες προμήθειες που θα λάβουν χώρα αφού τεθεί σε ισχύ. και έχω επίγνωση τότε θαύματα δεν γίνονται δεν μπορεί μόνο με την οδηγία να τα καταφέρουμε και φυσικά μπορεί να οργιάσει η φαντασία μας και να εντάξουμε κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες αλλά ίσως μπορούμε να ενεργήσουμε γενικότερα με κάποιο άλλο νομοθέτημα ούτως ώστε να προωθήσουμε τις προτάσεις μας. Επίσης, είναι πολύ θετικό όπως είπαν ε, κάποιοι συνάδελφοι ότι σας ε, αρέσει αυτή η προσέγγιση για την ε, οδηγία άφη σε σχέση με την παρούσα οδηγία Πάντως η αρχική μου ιδέα ήταν ότι αν έχουμε μια απαρίθμηση με τα επιλέξιμα ε, καύσιμα σε διάφορες διατάξεις ή ε, αυτό θα κάνει δυσχερέστερη την ε, επικαιροποίηση του νομοθετήματος οπότε ακριβώς είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτή η επικαιροποίηση αλλά να μην έχουμε από εδώ και από εκεί ε, τέτοιες ε, απαριθμίσεις, τέτοιες λίστες. Μάλλον αυτό δεν είναι τόσο χρήσιμο για την ε, βιομηχανία, γιατί μπερδεύονται με όλα αυτά. Πού να κάτσει κανείς όλα αυτά ταυτόχρονα να τα επικαιροποιήσει. Δεν είναι ρεαλιστικό. Γι' αυτό και διάλεξα να επισυνάψω εδώ τον κατάλογο των επιλεξίμων καυσίμων της οδηγίας ΣΑΦΗ πολύ θετικό όλο αυτό που είπατε όλοι, μάλλον όλοι για την ε, τεχνική ουδετερότητα. Ίσως όχι πράσινη, αλλά τι να κάνουμε. Σας άρεσε, αυτό είναι σημαντικό για όλους σας. Ωραία. Ναι, ναι, γνωρίζω την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν με έχετε πείσει όσον αφορά το ότι δεν έχετε αποδείξει αυτό που λέτε. Ε, γι' αυτό και εγώ έκανα κάποιες ε, μικρές αλλαγές. Ε, ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις τροπολογίες σας. Ε, εμείς ευχαριστούμε κύριε Ντελή. Σας υπενθυμίζω ότι η κατάθεση τροπολογιών είναι μέχρι τις 7 Ιουνίου στις 2 η ώρα. Αυτά. Αν είναι κάτι άλλο, ε, τότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ε, Δευτέρα 4 ε, Ιουνίου η Στάς 4. Με ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα συνεδρίαση.